Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε όλο και πιο ανησυχητικές και τραγικές ειδήσει από τη Μεσόγειο. Την Κυριακή, μετά από ένα ναυάγιο, υπάρχουν πάνω από 400 αγρόουμενοι από τις ακτές της Λιβύης, μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι, πολλά νέα άτομα και πολλά ανήλικα παιδιά. Υπάρχει ο φόβος ότι το μεγαλύτερο μέρος ε, των ατόμων αυτών έχει πνιγεί. Θα είναι μία από τις χειρότερες <laughs> τραγωδίες που εμπλέκουν πρόσφυγες από τον Οκτώβριο του 2014. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι σκέψεις μας στρέφονται προς τα θύματα και προς τις οικογένειές τους. θέλω να τονίσω και πάλι το πολύ δύσκολο ρόλο των δυνάμεων διάσωσης που εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες για να διασώσουν όσους μπορούν. Αυτές οι τραγωδίες μας αφήνουν άφωνους και μας υπενθυμίζουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση σε χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη και σε άλλες χώρες της Μεσογείου από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες στην Ελλάδα πρέπει κατεπηγόντως να δώσουμε πολιτικές λύσεις για τις χώρες αυτές. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα οι Ιταλοί διασώστες έχουν διασώσει 6.000 άτομα στη θάλασσα. Τα ε, ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα είναι τα πιο θανατηφόρα σύνορα στον κόσμο. Παρά από τις χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν από, διασχίζοντας τη Μεσόγειο στην Ευρώπη έχουν χάσει τη ζωή τους. Θα πρέπει να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα αυτά. Αλλά δεν μπορώ να πω αυτά που λέω χωρίς να σας υπενθυμίσω το ίδιο. Στις 17 Οκτωβρίου 13 βρισκόμουν ήδη σε αυτή την ίδια θέση και είχα ζητήσει ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Λαμπεδούσας. 15 Σεπτεμβρίου 2014 πάλι σας είχα καλέσει για ένα λεπτό συγγύηση για 200 πρόσφυγες που πνίγηκαν. Το Φεβρουάριο του 2015 πάλι για 300 μετανάστες που πνίγηκαν. Και σήμερα πάλι βρίσκομαι ενώπιόν σας και σας ζητώ και πάλι ένα λεπτό συγγύηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας τιμά να συνεχίζουμε μονάχα με λεπτά σιγής για τα εκατοντάδες θύματα χωρίς στην πράξη να μην αλλάζει τίποτα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό η έκκληση αυτή δεν αφορά μοναχα εμάς και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφορά κυρίως και απευθύνεται κυρίως στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπλέκει την ευθύνη τους για τη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, για να έχουμε καλύτερη προστασία των προσφύγων, αλλά και για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα αίτια αυτού του μεταναστευτικού ρεύματος. Τα κράτη που έχουν αστοχήσει τα αποτυχημένα κράτη στον περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αίτιο αυτού του μεταναστευτικού ρεύματος. Πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, αλλά είναι και στη δική μας ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε με εντατικό και ουσιαστικό τρόπο τα αίτια αυτής της μαζικής μετανάστευσης. Προσθέτω και την ε, τρομερή ε, επίθεση της Δευτέρας Απριλίου της Al-Shabaab στο Πανεπιστήμιο Λαρίσα στο βορρά της ε, όπου έχασαν τη ζωή τους 180 αθώοι φοιτητέ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τρομοκρατική αυτή οργάνωση με τέτοιο ομό και βίαιο τρόπο διαλέγει σε θύματα της αθώα άτομα. Αυτό μας έχει συγκλονίσει, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει γίνει κατά συρροή και επανάληψη και κυρίως εναντίον ατόμων χριστιανικής θρησκευτικής πίσης. Θα πρέπει και εδώ να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των ε, θυμάτων. Και εύχομαι στα άτομα που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς να αποθεραπευτούν το ταχύτερο να αποκατασταθεί η υγεία τους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγώνας κατά της νομοκρατίας δεν είναι μόνο αγώνας κατά μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι και ένας αγώνας για την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας. Είναι και η βάση, το θεμέλιο της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Για όλα αυτά τα θύματα λοιπόν σας ζητώ να σηκωθείτε και να κρατήσετε ένα λεπτό υγεία. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Μου ζητήθηκε κυρίε και κύριοι. Έχω κάτι χαρτιά. Και θα το πράξω μετά την στιγμή σιγής να σας υπενθυμίσω ότι στο Γιαρμούκ, στον καταβλισμό προσφύγων, στην Δαμασκό, όπου εδώ και δύο χρόνια βρίσκονται 18.000 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, είναι αποκλεισμένοι εκεί, φυλακισμένοι ουσιαστικά. Η κατάσταση η ανθρωπιστική στον θύλακο αυτό είναι ικτρή. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων είναι απόλυτα απομονωμένοι από τον κόσμο. Έχουν έλλειψη τροφίμων, νερού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και εκεί τώρα βρίσκονται τα στατέματα του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους που κρατούν αυτούς τους πρόσφυγες ως ε, όμοιρους, ως ανθρώπινες ασπίδες. Και γι' αυτό το λόγο ότι αυτό φυσικά δεν μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος πιστεύω ότι μπορώ να εκφράσω την άποψη όλων σας με το να κάνω μια έκκληση προς τους ένοπλους να φυστούν τη ζωή και τη ακαιρεότητα των γυναικών και των παιδιών στο Γιαρμούκ. Η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο Γιαρμούκ και να μπορέσει να εξασφαλίσει τα βασικά αγαθά στους αποκλεισμένους στο θύλακο του Γιαρμούκ. Η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή είναι αυτή που έχει επιληφθεί περισσότερο για το θέμα αυτό και έχει υποστηριχθεί μαζικά οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι και εσείς συμμερίζετε την άποψη ότι και η ούρα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από όλους μας και σε μία από τις μεταγενέστερες συνεδριάσεις μας θα πρέπει πάλι να κάνουμε και ενός λεπτού συγγύης για τα, τις ε, κατοντάδες θυμάτων στο Γιαρμούκ. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσουμε για χιλιάδες. Παρακαλώ όλους λοιπόν και αυτούς οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν πίεση σε, στους διεθνείς οργανισμούς, στις κυβερνήσεις τους μάλλον, να βοηθήσουν τους διεθνείς οργανισμούς στο έργο τους.